Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Άρχεται εκ νέου συνεδρίαση, κυρίε και κύριοι. Έχει μου μοιραστεί τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση και σα παρακαλώ να μου δηλώσετε αν υπάρχουν αντιρρήσει. Αν δεν υπάρχουν, εγκρίνονται τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη έχει τώρα πέντε ψηφίσματα για το Ιράν, για τη Σιρήνα Μπαντή.